Herr Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie bitten. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Es sich zu... Können Sie mal mit dem Klopfen aufhören, bitte. Παρακαλώ σταματήστε λίγο το, το θόρυβο. Ο Φράνσις Βούρτς ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς πρέπει να σας ενημερώσω